δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μαρία Τσέκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την βδομάδα του Πάσχα των ε, Ορθοδόξων στην Αίγυπτο δολοφονήθηκαν 10 κόπτες σε αυτή τη χώρα. Και βέβαιω, αν και το περιστατικό αυτό αφορούσε τους κόπτες, πρέπει να προστατεύουμε κάθε θρησκευτική μειονότητα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η βία και βεβαίω πρέπει να προστατεύσουμε τη θρησκευτική ελευθερία, αλλά και την ελευθερία από την θρησκεία και θα πρέπει οι διαφορές να λύνονται με ανοιχτό διάλογο. Και σε μια κοινωνία βεβαίω θα πρέπει οι ελευθερίες αυτές να είναι εγγυημένες. Μια ανοιχτή κοινωνία μπορεί να υπάρξει μόνο όταν η σχέση κράτους και εκκλησίας αναφέρεται στο Σύνταγμα. Τα μέτρα ασφαλείας δεν μπορούν να είναι τα αυτά τα οποία ισχύουν σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Και όμως τα τελευταία 28 χρόνια η Αίγυπτος είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η ανοιχτή συζήτηση ίσως είναι το πιο ισχυρό μέσο κατά του εξτρεμισμού, οπότε η ελευθερία έκφρασης στο ίντερνετ και εκτός μπορεί να μειώσει τις εντάσεις στην κοινωνία. Γι' αυτό είναι δύσκολο να αντιληφθούμε και να δεχτούμε το ότι γύρω στους 30 ακτιβιστές, πολιτικές και bloggers συνελήφθησαν ενώ ταξίδευαν στην πόλη του Ναγκαχαμάντι για να εκφράσουν τα συλληπιτήριά τους σε όσους δολοφονήθηκαν κατά την διάρκεια αυτών των επεισοδίων και πλέον έχουμε την ίδια συμπεριφορά που ακολουθείται μόνιμος από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Κάτι δεν πάει καλά όταν αντιμετωπίζουν κάποιους ως εγκληματίες μόνο και μόνο επειδή πάνε να εκφράσουν αλληλεγγύη με συμπατριώτες τους. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το επιχείρημα της δημόσιας τάξης υφίσταται κατάχρηση. Από το 2008 δεν μπορούν να πάρουν ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή οι Αιγύπτιοι, αλλά τώρα έχουν και άλλους κανόνες. Για να συνδεθεί κανείς στο ασύρματο ίντερνετ πρέπει να δώσει email και το συνθηματικό του. Οπότε η κυβέρνηση ελέγχει όλους τους χρήστες. Επίσης υπάρχει νόμος για τη ρύθμιση του διαδικτύου που προβλέπει φυλάκιση εάν κάποιος δημοσιεύσει περιεχόμενο χωρίς έγκριση της κυβέρνησης. Και όμως η κυβέρνηση λέει πως υπάρχει εγγύηση της ελευθερίας έκφρασης και κάθε άτομο είναι ελεύθερο να εκφράσει την άποψή του με οποιονδήποτε τρόπο εντός των ορίων του νόμου. Η αυτοκριτική και η επικοδομητική κριτική βεβαίως αποτελεί την βάση για την εθνική ασφάλεια. Θα ήθελα να ζητήσω από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση να μην εφαρμόσει τους νόμους εκτάκτης ανάγκης. Πρέπει να υπάρξει μια σωστή απάντηση στα εγκλήματα αυτά, δεν πρέπει όμως να καταπιεστεί όλος ο πληθυσμός με νόμους που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση. Μόνο όταν είναι όλα τα στρώματα του πληθυσμού ελεύθερα θα υπάρχει ανοιχτή κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν η Αίγυπτος να οδηγήσει πολύ στην ελευθερία και η Ευρώπη να την βοηθήσει. Σας ευχαριστώ κυρία Σάκε. Ο κύριος Προβέρα έχει τώρα τον λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ψήφισμα το οποίο παρουσίασα ξεκινάει από κάποια τραγικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν πρόσφατα στην ε, ε, Αίγυπτο και σε άλλα μέρη του κόσμου, χθε ας πούμε στην Ιγυρία, έτσι ώστε να ε, δείξει σε ολόκληρο τον κόσμο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την απαράδεκτη κατάσταση όσον αφορά διωγμούς και δολοφονίες μελών της κοινότητας. Δεν πρόκειται για ψήφισμα κατά της Αιγυπτιακής κυβέρνηση, η οποία έπραξε τα πάντα έτσι ώστε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη ε, οι ε, υπεύθυνοι αλλά πρόκειται για ένα ανησυχητικό και ευρύ φαινόμενο ε, Στου, ανάμεσα στο Βιετνάμ, τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα, το Ιράν, τη Μαλαισία, την Ιγυρία για να, μην, για να αναφέρω μόνο ορισμένες χώρες διαπιστώνουμε ανησυχητικά φαινόμενα διώξεων κατά των χριστιανικών κοινοτήτων που φτάνουν μέχρι τις Βεβαίω, τα πρέπει όλοι να δεσμευτούν έτσι ώστε να αλλάξει αυτό το κλίμα ε, θρησκευτικού μίσους το οποίο διαρκώς εξαπλούται και έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα. Η Ευρώπη γνωρίζει πάρα πολύ καλά την τραγωδία των πολέμων που για πολλούς αιώνες αντιπαρέθεσαν καθολικού ε, και διαμαρτυρόμενους, χωρίς να μιλήσουμε βεβαίω για το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Ακριβώς λόγω της ιστορίας της ε, η Ευρώπη θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Μία άλλη ε, πρωτοβουλία θα μπορούσε να αφορά τον έλεγχο των εθνικών νομοθεσιών, στα πλαίσια των οποίων βλέπουμε νόμου που από τη φύση του οθούν στην δίωξη των χριστιανών ή οποιονδήποτε άλλο χριστιανικό ε, μειονοτήτων. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους ε, μη κυβερνητικού οργανισμούς που μπορούν να μας βοηθήσουν στο σχέδιο αυτό. Και βεβαίως θα πρέπει να λάβει χώρα τέλος αυτή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάριο Μάουρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η θρησκευτική ελευθερία ε, αποτελεί θέμα αυτού του ψηφίσματος. Ε, καθόλου δεν πρόκειται εδώ για μία σταυροφορία όσον αφορά ε, την <clears throat> ταυτότητα κάποιων ανθρώπων. Αλλά αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο πεθαίνουν γιατί πιστεύουν στο Χριστό, γιατί πιστεύουν στο χριστιανισμό. Δηλαδή γιατί ζουν σε μία χώρα όπου κάποιοι τους λένε πρέπει να πεθάνεις γιατί πιστεύεις κάτι διαφορετικό διαφορετικό από Γι' αυτό ακριβώ το ζήτημα τούτο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τρόπο σταθερό και συγκεκριμένο σαν ε, ε, διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητούμε από την είπατε εκπρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αναλυφθούν άμεσα πρωτοβουλίες ε, οι οποίες ε, θα οδηγήσουν σε διάλογο μεταξύ όλων των κοινοτήτων και βεβαίως ε, που θα μπορέσουν να σταματήσουν και να αποδυναμώσουν εν τη γενέση οποιαδήποτε τέτοιου είδους κινήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βερονίκ Ντεκεζέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αυτά που συνέβησαν ε, στην Αίγυπτο θα μπορούσαν να είχαν συμβεί και αλλού. Ένα αυτοκίνητο ε, περνάει έξω από ένα ε, ναό <clears throat> και ξεκινούν οι πυροβολισμοί οι οποίοι έχουν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ανθρώπων. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Αιγύπτου αποφάσισε ότι οι τρεις υπεύθυνοι για τα συμβάντα σε αυτήν την περιοχή της Αιγύπτου θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να προσαχθούν ε, τις πόλεις ε, Ναγκά Χαμαντή, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσαχθούν στο έκτο δικαστήριο κρατικής ασφάλειας για φόνο εκπρομελέτης. Αυτά, αυτή είναι όντως μια καλή αντιμετώπιση. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνομαι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο η υπάρχει μία αναμόχλευση των ε, παθών. Ε, ε, σε ολόκληρο τον κόσμο βλέπουμε ότι διαπράττονται αδικήματα, εγκλήματα κατά μειονοτήτων, θρησκευτικών, πολιτικών κτλ. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες φυλακίζονται και διώκονται γυναίκες οι οποίες αρνούνται να υποταχθούν σε δόγματα, δοξασίες και πρακτικές οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ξεχαστεί από χρόνια. Εγώ ε, σαν υπέρμαχος του κοσμικού κράτους δεν είναι δυνατό να δεχτώ ε, όλα όσα συμβαίνουν στην Μαλαισία σε άλλες χώρες του κόσμου. Ένα κοσμικό κράτος το οποίο θα είναι κοσμικό σε όλες του τις ε, διαρθρώσεις είναι η μόνη δυνατότητα προστασίας των πολιτών και ευνόησης του διαλόγου μεταξύ των κοινοτήτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεκεζέρ. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ο κύριος Λεγκούρκο. Mr. President, Madam Commissioner. Κύριε, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι πληροφορίες για τη βία κατά των χριστιανών στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου. Τρία σημεία θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα οι χριστιανοί έχουν γίνει θύματα βίας σε πολλές χώρες, όχι μόνο σε αυτές. Δεύτερον, οι χριστιανοί έχουν γίνει η πιο διοκόμενη θρησκεία στον κόσμο. Τα νούμερα είναι εκπληκτικά, είναι στα εκατομμύρια, όχι στις ε, χιλιάδες, το ύψος των περιπτώσεων. Τρίτον, η αντίδραση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, κυβερνήσεων και της Ένωσης ήταν μέχρι στιγμής μη ικανοποιητική. Δειλή, ψοφοδεής, και πολιτικά ορθή ή καμία αντίδραση. Πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά, αλλιώς όσοι διώκουν τους χριστιανούς θα θεωρούν ότι έχουν και την σιωπηρή μας ανοχή. Το θέλουμε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Λεγούτκο. Τον λόγο για ένα μισή λεπτό έχει η κυρία Χάουτελα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Χάουτελα. Είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι έχουμε τόσες συγκρούσεις στον σύγχρονο κόσμο που προκαλούνται από θρησκευτικέ διαφορές. Οπότε, τελικά έχουμε πολλούς φονταμεταλισμούς. Και όχι μόνο τον μομεθανικό φανατισμό, για ίσως είναι ο βουδισμός που δεν δημιουργεί τέτοιου ακραίες τάσεις. Κάθε φορά επομένω ασχολείται το Κοινοβούλιο με τέτοιου είδου ε, ε, βία, γεγονότα βία συγκρούσεων μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων. Πάντω, χθε μόλι μάθαμε ότι 33 αγωνιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν όταν διαδήλωσαν υπέρ των χριστιανών που αναφέρονται στο ψήφισμα. Και θα πρέπει να στείλουμε μήνυμα προς τις ε, Αιγυπτιακές αρχές. Δεν είναι δυνατόν να εμποδίζονται αυτοί που θέλουν να υπερασπιστούν κάποιον άλλο. Δεν θα πρέπει να φυλακίζονται τέτοια πρόσωπα που υπερασπίζονται τα δικαιώματα κάποιου άλλου. Αυτό έγινε με αυτού τους 33 ε, ε, οι οποίοι τελικά σαν απάνθρωποι μεταχείριση κατά την κράτηση. Στο μέλλον ελπίζουμε το κοινοβούλιο να προσέχει τέτοιου είδου ε, ζητήματα που δημιουργούνται και με άλλε τρει και όχι μόνο με προβλήματα των χριστιανών. Και τώρα, εκπρόσωπο των πολιτικών ομάδων για το Λαϊκό Κόμμα. Για ένα λεπτό, κύριο Πόσελτ κύριε Πρόεδρε, η Τινησία, η Αίγυπτος και η Μαλαισία έχουν μεγάλη παράδοση ανεκτικότητας. Ο ιδρυτής της Μαλαισίας, ο Τούνκο Αντουλαχμάν ή ο πρόεδρος Σαντάτ, νομίζω μπορούν να ε, μας υπενθυμίσουν εδώ πέρα ακριβώς αυτή την Μάγνα Χάρτα των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων. Γι' αυτό νομίζω πως πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το ψήσμα κατά δίκης των ε, επιθέσεων αυτών. Και γι' αυτό έχουμε την ευθύνη εμείς ως κατά πλειοψηφία χριστιανική Ήπειρος να τοποθετηθούμε. Αλλά είναι βεβαίως πως είναι αυτονόητο πως πρέπει να υπάρξει σκεφτική ελευθερία και θέλω να ευχαριστήσω τον βασιλιά της ε, Μαλαισίας για το ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό έλαβε θέση ήδη από τις 9 Ιανουαρίου και ελπίζω να έχουν επιτυχία στον αγώνα τους καταπολέμησης της θρησκευτική μη ανεκτικότητας κάτι το οποίο πρέπει να βοηθήσουμε και στις τρεις αυτές χώρες Αίγυπτο, Μαλαισία και την Ισία, ειδικά στη συνεργασία μας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές για ένα λεπτό ο κύριος Φαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικό κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ελευθερία άσκησης σκεφτικής των σκεφτικών καθηκόντων. Βλέπουμε όμως ε, πως αυτό εμποδίζεται σε χώρες ε, όσον αφορά χριστιανούς, σε μουσουλμανικές χώρες οι κόπτες στην ε, Αίγυπτο και οι Ιουδαίοι και ε, άλλες ε, χριστιανικά δόγματα καταπιέζονται. Αυτό επίσης αναφέρεται η θρησκεία τους και στα έγγραφα ταυτότητας και στα λοιπά. Τα τελευταία λοιπόν δέκα με 20 χρόνια αυξηθεί πάρα πολύ η πίεση εναντίον των κοπτών. Έχουν υπάρξει πάνω από 100 επιθέσεις με χιλιάδες θύματα και θεωρώ πως δεν υπήρξε σοβαρή αντίδραση της Αιγυπτιακής ε, κυβέρνηση συνελήφθησαν τρία άτομα, αλλά δεν υπήρξε καμία σοβαρή διερεύνηση. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε την κυβέρνηση για να αλλάξει πορεία και αν δεν το κάνει το Κάιρο θα πρέπει αυτό να έχει επιπτώσεις στις διμερείς μα σχέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά έχει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Χίγγινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε όλοι όσοι παλεύουν για δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερία τη έκφραση δεν μπορούν παρά να καταδικάσουν τις δολοφονίες αυτές των ε, χριστιανών στην ε, Αίγυπτο και την πυρπόληση των εκκλησιών στη Μαλαισία. Και στην Ευρώπη βέβαια θα πρέπει να προστατεύονται τι θρησκευτικέ μειονότητε. Ε, στην Μαλαισία πάντοτε χρησιμοποιούσαν αυτό το διέρη και βασίλευε οι, οι ελίτες της εξουσίας. Και το κάνουν όλα αυτά ενώ διακηρύσουν ότι προστατεύουν όλες τις μειονότητες. Όμως βάζουν να αντιπαρατεθεί μία μειονότητα εναντί της άλλης ή μία κοινότητα εναντί της άλλης για να διακυβερνήσουν καλύτερα. Στην η Ασία είναι η πιο άνηση κοινωνία. Εκμετάλλευση των εργαζόμενων, ε, καταπίεση των συνδικαλιστών. Επίσης, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η κατάσταση ε, σε, σε Αίγυπτο και Μαλαισία είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι η ανάπτυξη της οικονομική πάει με χέρι με τη δημοκρατική μεταρρύθμιση. Ευχαριστούμε κύριε Χίγκη, το πρώτος και τώρα. Στους μη γεγραμμένους, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριο. Φαντερστούπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χτες ξεκίνησε στην Ολλανδία μια φρικτή πολιτική δίκη κατά του Προέδρου μας, του Χέρτ Βίλτερς, ως ε, Ολλανδός βουλευτής του Ολλανδικού Κοινοβουλίου διώκεται για την γνώμη του από τις ελίτ ακριβώς για το ότι προειδοποιεί την Ευρώπη και τον κόσμο για τη φασιστική ιδεολογία του Ισλάμ κύριε Πρόεδρο, ο εξισλαμισμός της Ολλανδίας και της ε, Ευρώπης απειλεί την Ιουδεοχριστιανική, τον Ιουδεοχριστιανικό πολιτισμό. Και το τσουνάμι του εξισλαμισμού θα έρθει. Γι' αυτό το κόμμα μας υπερασπίζεται τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα και στην Αίγυπτο και στη Μαλισσία και σε πάρα πολλά άλλα μέρη του κόσμου αποτελούν απλό επακόλουθο της φασιστικής ιδεολογίας του Ισλάμ. Οι μουσουλμανικές χώρες στις οποίες κατά σύστημα καταπιέζονται οι χριστιανοί πρέπει επιτέλους να δουν πως αυτά τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Έχουν τις ρίζες της σε μη ιδεολογία η οποία είναι μη ανεκτική. Είναι τρομακτικά γεγονότα τα οποία δεν πρέπει να συμβούν ποτέ στην Ευρώπη. Γι' αυτό σας καλώ να παλέψουμε όλοι μαζί με το κόμμα μας για να αποφευθεί ο εξισλαμισμός της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο πρώτος, ευχαριστούμε κύριε Φαντεστούρ και τώρα. Οι επόμενοι βουλευτέ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ο κύριος Κάτσμουρεκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Συχνά στο Κοινοβούλιο ε, συζητούμε για διάφορες ε, φοβίες, ξενοφοβία ε, κτλ. Αλλά οι φοβίες τις οποίες συζητούμε, στις φοβίες μάλλον που συζητούμε, ξεχνούμε να αναφέρουμε την χριστιανοφοβία. Αυτή η φοβία λοιπόν είναι μια φοβία η οποία έχει οδηγήσει σε πολύ αρνητικά, βλέπε τραγικά αποτελέσματα και συνέπειες ε, και βεβαίως καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, βεβαίως εμείς θα πρέπει, χωρίς να ξεκινήσουμε σταυροφορία, να υπεραμεινθούμε των δικαιωμάτων των ε, χριστιανών, γιατί φυσικά η Ευρώπη μεταξύ άλλων βασίζεται και στον πυλώνα που λέγεται ε, ελευθερία έκφρασης και ελευθερία ε, θρησκευτική πίστης. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασμάρεκ. Για ένα λεπτό ο κύριος Σιμάνσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα δικαίωμα το οποίο περιλαμβάνεται εδώ και 50 χρόνια στις διεθνείς συνθήκες. Όμως τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ένα κύμα θρησκευτικού μίσους εναντίον των ε, χριστιανών ε, και ε, τα προηγούμενα χρόνια αυτό το κύμα ξεκινούσε από τους κομμουνιστές. Τώρα ξεκινάει από τους φανατικούς φανατικούς ε, ε, Ισλαμιστές. Γνωρίζομαι ότι ειδικά ε, στα μουσουλμανικά κράτη οι ακραίες θέσεις λαμβάνονται και δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων στο όνομα της χριστιανοφοβίας ή της χριστοφοβίας διαπράττονται εγκλήματα και βεβαίως θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιμάνς και ο κύριος Σόνικ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Συμφωνώ με τον κύριο Προβέρα. Θα πρέπει να συντάξουμε μια έκθεση σε σχέση με τις θρησκευτικές ε, Σε αυτό αναφέρθηκα και εγώ, αλλά και ο κύριος Μάουρο σε σχέση με μια τέτοια έκθεση όσον αφορά τις ε, χριστιανικές μειονότητες. Τελικά όμως δεν βρήκαμε υποστήριξη στην πρότασή μας. Θα πρέπει περίφραστα να τοποθετηθούμε υπέρ των αδελφών χριστιανών. Κάθε φορά που υφίστανται πίεση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματά τους, θα θρησκευτικά. Με μεγάλη προσοχή μελέτησα την ε, επιστολή του που απευθύνθηκε στον ε, πρόεδρο Μπούζεκ. Βεβαίω και πρέπει να γίνουν σεβαστά αυτά τα σκεφτεία δικαιώματα. Ε, ο πρόεδρος. Κύριε Σόνικ, ευχαριστούμε. Τσαρνέτσκι, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το θέμα δεν είναι μόνο η Αίγυπτος και η Μαλαισία, είναι και το Σουδάν και η Νιγηρία και άλλες χώρες στην Αφρική και κάποιες χώρες στην Ασία. Και κάποιες κοινωνίες μεταχειρίζονται τους χριστιανούς σαν άτομα ανεπιθύμητα ή εχθρούς. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμείς προσπαθούμε να αγνοήσουμε το πρόβλημα. Είναι όμως ένα πραγματικό πρόβλημα. Στην χριστιανική Ευρώπη έχουμε την κληρονομιά μας, οπότε πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας, να παραδεχτούμε ότι είμαστε ένοχοι. Έχει υποθεί πως ε, έχουμε υποπέσει σε παραλήψεις. Πράγματι, πριν από λίγες εβδομάδες καταδικάσαμε τις επιθέσεις ε, και τις διώξεις της μουσουλμανικής κοινότητας στην Κίνα αλλά κάποιες πολιτικές ομάδες μετά ήταν κατά τροπολογιών που τόνιζαν ότι και οι χριστιανοί διώκονται στην Κίνα. Οπότε δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε μόνο μερικές θρησκείες και άλλες όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κόριολα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ ακούσαμε κάποιες ανησυχητικές πληροφορίες από διάφορες πηγές για εγκλήματα κατά χριστιανών και στην Αίγυπτο και στην Μαλαισία. Όσον αφορά τη Μαλαισία θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για τις επιθέσεις της Εκκλησίας σε μια χώρα που παραδοσιακά ήταν ανεκτική. Κατόπιν θα ήθελα να τονίσω το εξαιρετικό έργο Ισλαμικών μη για να αυξηθεί η ανεκτικότητα Επίσης, το ότι έγιναν δηλώσεις ε, από τον Πρωθυπουργό για να απαγορευτεί η χρήση της λέξης Αλλάχ οδήγησαν σε αυτά τα επεισόδια και βεβαίως οι Ισλαμικές ΜΚΟ καταδίκασαν αυτή την στάση. Πρέπει να συμπεριληφθούν αυτά ε, και στο ψήφισμά μας. Δεν πρέπει να ευχαριστήσουμε τις μουσουλμανικές ΜΚΟ για τις δηλώσεις τους αυτές είναι εξίσου σημαντικό να σημειώσουμε βεβαίως και τα αρνητικά και τα θετικά βήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Μποντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι πράξεις ε, φανατικών εγκληματιών που δολοφόνησαν χριστιανούς δεν μπορούν να ε, χαρακτηρίσουν μια χώρα ολόκληρη και την κυβέρνησή της. Θα ήταν άδικο να θεωρήσουμε υπεύθυνους την Αίγυπτο, την Αιγυπτική κυβέρνηση και τους Αιγυπτίους για αυτήν την απεχθή πράξη, οι ε, υπεύθυνοι της οποίας πρόκειται να δικαστούν. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε αμάλγαμα ανάμεσα σε ορισμένους φανατικούς και μια ολόκληρη χώρα και έναν ολόκληρο πληθυσμό. Βεβαίως, ανάμεσα στους χριστιανούς κόπτες της Αιγύπτου ε, και τους μουσουλμάνους της Αιγύπτου ενδεχομένως υπάρχουν κάποια προβλήματα. Απ' την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε θέσεις οι οποίες θεωρούν ότι οι χριστιανοί της Αιγύπτου είναι κατάσκοποι της δύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τόκες. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Μάθαμε πρόσφατα πως πριν από λίγες ημέρες οι Αιγυπτιακές αρχές συνέλαβαν υπερασιστές ε, νομικούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τους πήγαν στον Καμαντή ε, όπου είχαν πάει για να υπερασπιστούν τους κόπτες ε, ε, εκπρόσωποι των οποίων δολοφονήθηκαν τα Χριστούγεννα. Οι Αιγυπτιακές ε, αρχές ε, προσπαθούν να πούν πως δεν ήταν τίποτα τόσο σπουδαίο οι ε, πράξευτες κατά των μειονοτήτων και δεν τους επιτρέπουν και να αμυνθούν. Καταδίκασαν και οι ΙΠΑ αυτές τις επιθέσεις. Γνωρίζουμε πως οι κόπτες είναι αρχαίοι κάτοικοι της Αιγύπτου. Εδώ και χιλιάδες χρόνια υφίστανται καταπίεση. Γι' αυτό πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα να τους προστατεύσει αποφασιστικά. Ευχαριστώ. Κύριε ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν ζητήσει το λόγο για τη διαδικασία ΚΑΤΣ ΔΙΑΕ. Στις 12 θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία. Εκ των 8, 4 μπορούμε να λάβουν το λόγο. Ένας από κάθε πολιτική ομάδα, από τις πολιτικές ομάδες που ανήκουν αυτοί που ζήτησαν το λόγο. Για ένα λεπτό πρώτη, έχει το λόγο κυρία Ζαμπόρσκα. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους καταδίκασαν την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών όπως είχε γίνει και το 2007 και το 2008. Δεν ξέρω τώρα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται πραγματικά να υπερασπιστεί συνεπώς τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί ακούμε συνέχεια τα ίδια παράπονα, αλλά δεν ακούμε εδώ πέρα κάποια υπεράσπιση των χριστιανών που δολοφονούνται, που τους κλείνουν τις εκκλησίες. Πράγματα που συμβαίνουν και στην Ινδία, στην Κίνα, στο Πακιστάν και σε πολλές άλλες χώρες. Οι χριστιανοί απειλούνται από ακραία ρεύματα. Αυτό ισχύει για όλους. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε όλους τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους τους ευρωβουλευτές να συνεισφέρουν σε ένα καλύτερο διαλογό για την ανεκτικότητα και για καλύτερη συνύπαρξη. Σας ευχαριστώ κύριε Ρεπού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση στην Αίγυπτο γιατί σχετίζεται με ζητήματα ιστορικά, εθνοτικά και άλλα. Οι κόπτες είναι μια πάρα πολύ σημαντική μειονότητα, είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια, 10% του πληθυσμού είναι υπερήφανοι για το ότι είναι κόπτες και για την παράδοσή τους Γι' αυτό ακριβώς η επίθεση αυτή ήταν εξαιρετικά βίαιη και προμελετημένη το γεγονός ότι πολλές γυναίκες ε, που ήταν κόπτες ξαναγκάστηκαν να αλλάξουν ε, θρησκεία και βιάστηκαν μεταξύ ναι, ναι. άλλων ε, είναι τραγικό και είναι θλιβερό αυτό το παράδειγμα που δίνεται και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε τον διάλογο μεταξύ των θρησκείων. Ευχαριστώ κύριε Ρέπο, κύριε Σφάγερ. Κύριε Πρόεδρε, κάθε φορά που έχουμε κάποια δολοφονία, κάποια ανθρωποκτονία που έχει ελαττήρια θρησκευτικά, τότε δεν ξέρει κανείς τι να πει. Θα πρέπει φυσικά να καταδικάσει τέτοιου πράξεις, αλλά αυτό δεν αρκεί. Να, άλλο ένα έγκλημα, το οποίο έγινε στην Μέση Ανατολή για αυτούς τους λόγους, όμως αυτό αντικατοπτρίζει, συγγνώμη, μία γενικότερη κατάσταση, ένα γενικότερο κλίμα, τότε δηλαδή δεν είναι σεβαστές οι θρησκευτικές ελευθερίες. Των μειονοτήτων βέβαια. Δεν υπάρχει επομένως ανεκτικότητα. έχουμε αυτή την πρόταση της ε, Άλντε, ούτως ώστε να συζητηθεί το πρόβλημα αυτό σε Αίγυπτο και Μαλαισία ε, θέλησαν χωριστή συζήτηση και εμεί αυτό το κάναμε γιατί θεωρήσαμε ότι θα πρέπει το κάθε θέμα να συζητείται χωριστά. Παρ' όλα αυτά όμω η Αίγυπτος δεν είναι η χειρότερη χώρα στον της του και των ελευθεριών. Το αντίθετο. Για ένα λεπτό κύριο Στάνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δυστυχώς το γενικότερο κλίμα στον μουσουλμανικό κόσμο είναι το να ενισχύεται η τζιχάντ, οι φανατικοί, ε, να χτυπιούνται οι χριστιανικές μειονότητες και όχι μόνο. Να, οι κόπτες σε μια παλαιότερες εκκλησίες. Στο Λονδίνο υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες τους. Ε, ήρθαν ε, κάποιοι ψηφοφοροι δικοί μου κόπτες και μου είπαν το τι γίνεται στην Αίγυπτο. Η μουσουλμανική αδελφότητα αυτά τα ενορχιστρώνει και παρά τις υποσχέσεις ε, του πρόεδρου Μουμπάρα και της κυβέρνησής του τα πράγματα πάνε στο χειρότερο έχουμε τους ε, χριστιανούς σε Συρία, σε Ιράκ, σε Παλαιστίνη ε, όλοι αυτοί χτυπιούνται τώρα βλέπουμε το ίδιο γίνεται και στην Μαλαισία το κοινοβούλιο νομίζω πάρα πολύ καιρό έχει να ασχοληθεί με την προστασία αυτών των μειονοτήτων οπότε νομίζω αυτό το ψήφισμα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό κύριε Τάνο ευχαριστούμε λίγο. πρόεδρος και Τελευταίο Αγορητή ο κύριο Μπάντεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι διώξει χριστιανών και άλλων μειονοτήτων σε Ισλαμικές χώρες είναι μόνιμο φαινόμενο, α πούμε στην Αίγυπτο, στην Μεσόγειο γενικότερα. Πάνω από 2.000 χρόνια ζουν χριστιανοί. Και παρόλα αυτά όμω φύσατε αυτέ όλε διώξεις γι' αυτό γιατί όλο ένα και πιο ισχυροί γίνονται οι φανατικοί, οι ακραίοι ε, οι Ισλαμικοί αυτοί οι Ισλαμοφασίστες και οπότε υφίσανται όλα αυτά οι μειονότητες ε, είναι κάτι όμως που τα ΜΜΕ στη Δύση μάλλον έχουν υποτιμήσει μάλλον θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος του τι γίνεται και γιατί γίνεται θα πρέπει να καταγγελθεί. Ποιο θα κάνει αυτά, δηλαδή φανατικοί μουσουλμάνοι. Και για ποιο λόγο το κάνουν, διότι γνωρίζει η άνθηση μια τέτοια ακραία ιδεολογία στον μουσουλμανικό κόσμο. Θα πρέπει δε να αυξηθεί η διπλωματική πίεση προ χώρε όπω ε, η Αίγυπτο, ώστε να σταματήσουν αυτέ οι αφόρητε διώξει. Κύριε Μπάτεν, σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα έχει το λόγο η Επίτροπο, η κυρία Κρού. Ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η Κομισιόν είναι σοκαρισμένη και θλίβεται βαθύτατα για τα περιστατικά στην Νότια Αίγυπτο και τον τραγικό θάνατο έξι κοπτών και ενός μουσουλμάνου αστυνομικού στην επίθεση αυτή. Είμαστε πεπισμένοι πως οι αρχές ανέλαβαν γρήγορα δράση για να βρουν τους υπόπτους κύριε Πρόεδρε, μια επισταμένη έρευνα θα στείλει οπωσδήποτε το μήνυμα πως η θρησκευτική βία δεν είναι αποδεκτή στην Αιγυπτιακή κοινωνία. Το Σύνταγμα της Αιγύπτου προβλέπει ε, θρησκευτική ελευθερία, όμως ακούμε παράπονα διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των κοπτών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων και στο χώρο εργασία και στα δικαστήρια. Και γνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι αλλάζουν θρησκεία και σπάζονται το χριστιανισμό όπως η Γκόρη Μοχαμετγάζη και τα προβλήματα που έχουν στα δικαστήρια. Φύγουμε αυτά τα ζητήματα στον πολιτικό διάλογο με την Αίγυπτο, αντιλαμβανόμαστε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια από τα παράπονα των κοπτών, π.χ. με το να μην καθυστερεί η άδεια οικοδόμησης και ανακαίνησης ναών και ζητούμε από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις ε, αιτίε ε, των θρησκευτικών εντάσεων στην κοινωνία και να σταματήσει κάθε διακριτική μεταχείριση των θρησκειών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ο βανδαλισμό εκκλησιών στη Μαλαισία μετά από μια απόφαση δικαστηρίου για τη χρήση τη λέξεω Αλλάχ προκαλεί σοβαρή ανησυχία η κυβέρνηση όπως και η αντιπολίτευση και το μαλισιακό Ισλαμικό κόμμα και 130 μουσουλμανικοί ΜΚΟ καταδίκασαν αυτές τις επιθέσεις. Η κυβέρνηση αύξησε τα μέτρα ασφαλείας στους ναούς και Επαναβίωσε την δεσμευσή της για να προστατεύσει την θρησκευτική αρμονία και ποικιλότητα. Το δε σύνταγμα της Μαλασίας αναφέρει πως το Ισλάμ είναι η θρησκεία της Ομοσπονδίας, αλλά επιτρέπεται εξάσκηση άλλων θρησκειών εν ειρήνη και αρμονία σε οποιοδήποτε τμήμα της χώρας. Ενθαρρύνουμε τις αρχές, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό έναν συνολικό διάλογο με όλα τα δόγματα για να προωθηθεί η κατανόηση, για να συνεχίσει η Μαλαισία την ειρηνική της ανάπτυξη εν και αρμονία. Και το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ πέρα έχει ιδιαίτερη ευθύνη για να εξηγήσει αντικειμενικά στους πολίτες το εν λόγω ζήτημα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταδικάζουμε όλες τις πράξεις μη ανεκτικότητας ε, κατά οποιοδήποτε για λόγους θρησκείας ή πεπιθήσεων. Δυστυχώς καμία χώρα δεν είναι πλήρω προστατευμένη από κάτι τέτοιο. Ζητάμε από όλε τι δημόσιες αρχές να προστατεύσει τι χριστιανικέ μειονότητε και του χριστιανού από την καταπίεση και τι διακρίσει και δίνουμε υψηλή προτεραιότητα στην ελευθερία, την θρησκευτική και την πεποίθηση και βεβαίω στείλουμε αυτό το ζήτημα στον διάλογο με τι χώρε αυτέ, με το να υποστηρίζουμε έργα ανθρώπινων δικαιωμάτων και με το να προωθούμε την θρησκευτική ελευθερία και στον ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Κλείνουμε το σημείο αυτό που θα, θα ψηφιστεί ε, μετά στις 12 δηλαδή. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Ιδίως ε, δε ε, θα αναφερθούμε στην περίπτωση του ε, Κινέζου Λίου Τσιάο Μπάο. Για, δύο, για δυόμιση λεπτά έχει τον λόγο η κυρία Βέμπερ.